Ε, περίπου δύο ώρες και τώρα θα μιλήσουμε για τις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου το άρθρο 135 του κανονισμού. Η συζήτηση πρώτη αφορά την κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στο Μαλάουι και σε άλλες αφρικανικές χώρες. Έχουμε ένα σύνολο συντακτών, οκτώ στο σύνολο για αυτό το ψήφισμα και ξεκινάμε δίνοντας το λόγο στην κυρία Μποντίλ Βαλέρο. Σας ευχαριστώ. Ένας άνθρωπος στις 20.000 στον κόσμο υποφέρει από το αλφινισμό και πολλοί εξ αυτών βρίσκονται, συγγνώμη, και πολύ ε, μεγάλη πλειοψηφία αυτών βρίσκονται στην Αφρική. 600 επιθέσεις δέχτηκαν αυτοί οι άνθρωποι σε 26 χώρες ε, τον περασμένο χρόνο γιατί ε, αυτοί χρησιμοποιούν μάλλον εκεί τα κάποια τμήματα του ανθρώπινου ε, σώματος αυτών των ε, ε, ανθρώπων Πρέπει λοιπόν να διωχθούν αυτά τα εγκλήματα και να προστατευτούν οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να δώσουν την μαρτυρία τους. Πρόκειται θέλουμε μια σοβαρή ε, απόφαση για αυτή τη σοβαρή απειλή για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα. Να υπάρξει ευαισθητοποίηση, να γίνουν εκστρατείε με στόχο την κοινή γνώμη που θα δουλεύει, που θα δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον αλφισμό γιατί πολλοί άνθρωποι πλήττονται από αυτή τη διπλή διάκριση Περισσότερη αστυνομική παρουσία, περισσότερη ενημέρωση και καταπολέμηση της στόχες και της διάκρισης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν περισσότερο από άλλες ομάδες ε, πληθυσμών. Tak, thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μαγέσο Ίσακ. Έτσι λέγεται το τελευταίο θύμα που γνωρίζουμε. Ένα αθώος νέος, ένα παιδάκι 12 ετών, που απήχθη, δολοφονήθηκε λόγω του ότι θεωρούν ότι τα μαλλιά του και το δέρμα του έχουν μαγικές δυνάμεις. Αυτό συμβαίνει. Τους τελευταίους εννέα μήνες το Μαλάουι ξανά ζει φρικτά εγκλήματα εις βάρος των ανθρώπων με αλφισμό. Πέρα από τη γνωστή διακριτική μεταχείριση και τα λοιπά, όλα αυτά είναι η κόρφη του παγόβουνου. Διαβάζουμε σε εκτές 600 άτομα που έχουν δολοφονηθεί. 21.000 άτομα στην Αφρική έχουν αλφισμό. Και πρέπει να φροντίσουμε και για τα δικά τους ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν επειδή έχουν διαφορετική όψη να τους δολοφονούν. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μακριά μας και στην Αφρική συμβαίνουν αυτά. Όχι. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε εν έτη 2017 να σταματήσει αυτή η δυσυδαιμονία. Πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση. Πρέπει οι εγκληματικές οργανώσεις που κάνουν εμπόριο των μελών αυτών των ανθρώπων να σταματήσουν. Γιατί, γιατί θεωρούν ότι τα ξανθά του μαλλιά έχουν μαγικέ δυνάμεις και δολοφονούν τα παιδιά με αλφισμό. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ, να φροντίσουμε ο καθένας πάνω σε αυτή τη γη, άσπρος, μαύρος, κίτρινος, να ε, έχει ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μιγγέλ Ουρμπάν Κρέσπο. Παρακαλώ. Ε, ο αριθμός των επιθέσεων, των εξαφανίσεων, όπως επίσης και των δολοφονιών στο Μαλάουι, στο, ε, στο Μπουρούντι. Τα τελευταία χρόνια 20 δολοφονίες και 115 έπεσαν θύματα αβίαιων επιθέσεων και φυσικά υπάρχουν και άγνωστες περιπτώσεις. Η κυβέρνηση του Μαλάουι θα πρέπει να πάρει νομικά και πολιτικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις αυτές οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαιτήσουν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών, της κοινότητας αυτής. Δεν μπορούμε να ζητάμε την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αφηρημένο τρόπο. Θα πρέπει εμείς να χρησιμοποιήσουμε τις ε, οικονομικές δυνατότητες ε, που έχουμε έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι καταστροφές. Η βία εις βάρος των ανθρώπων που υποφέρουν από αλφισμό δεν δείχνουν μόνο προκατάληψη, δείχνουν φτώχεια και απελπισία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρέσπο. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Κέλαμ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Επίτροπε, η... τα θύματα του αλφισμού στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ε, πολλαπλές διώξεις και διακρίσεις. 172 δολοφονήθηκαν πρόσφατα, υπάρχουν άλλες 300 επιθέσεις εις βάρος τους. Στο Μαλάουι έχει ξεκινήσει ε, φέτος μια νέα επίθεση εναντίον των ανθρώπων αυτών και τα δικαστήρια δεν μπορούν να προστατεύσουν την κοινότητα αυτή. Απευθύνουμε έκκληση στις αρχές του Μαλάουι να κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τους πολίτες ε, της χώρας αυτής. Θα πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις για την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια τους να ακολουθήσει το Μαλάουι τα θετικά παραδείγματα της Τανζανίας και της Μοζαμβίκης που βοήθησαν να συνειδητοποιηθεί το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Σοραγιά Πόστ. Ε, ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μιλήσω σου ειδικά. Συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, το κατεπήγον αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ να στήριξω. το πρόβλημα δηλαδή με τους αλφικούς στο Μαλάουι και άλλες χώρες της Αφρικής. Πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οι αλφικοί δολοφονούνται, υφίστανται καθημερινές διακρίσεις και ακόμη και οι δολοφονημένοι ακόμα δεν βρίσκουν ησυχία γιατί μετά ε, κατεργάζονται τα μέλη τους. Ε, οι γυναίκες και τα παιδιά είναι σε ακόμη χειρότερη θέση κόβουν τα μέλη τους και τα πουλάνε. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για την κατάσταση αυτή. Ζητάμε καλύτερη νομοθεσία και καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και περισσότερους πόρους για την αστυνομία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια εδώ πέρα. Χρειάζεται κάποιο σύστημα παρακολούθησης για να ξέρουμε το τι γίνεται. Και επίσης ε, υπάρχει ε, διαρθρωτικό πρόβλημα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων. Δεν μπορεί να αφήσουμε ανθρώπους να πεθαίνουν λόγω του χρώματος, του δέρματος τους. Είναι 2017. Χρειάζεται προστασία για όλους τους ανθρώπους της ε, χώρες αυτές και πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κύριο Στάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, η μοίρα των αλφικών στο Μαλάουι είναι τραγική και θυμάμαι την συζήτηση που κάναμε πριν από μία δεκαετία για την Τανζανία. Υπάρχει, υπάρχουν φρικτές δολοφονίες αλφικών ε, για διαμελισμό τους και σε χώρες εκτός του Μαλάουι, ειδικά παιδιών σε άλλες, ε, ε, χώρες, άλλες είναι το Μπουρούντι, η Μοζαμβίκη, η Κένια, η Νιγηρία και η Ζάμπια. Ήδη η κοινότητα αυτή κινδυνεύει ε, λόγω του ότι ζουν στους τροπικούς και κινδυνεύουν περισσότερο από καρκίνο του δέρματος. Αλλά τώρα πλέον κινδυνεύουν γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη η οποία ομοιάζει με μεσαιωνική μαγεία. Επίσης καλωσορίζω την ε, υιοθέτηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης 2017-2021 από την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ. Ένα συγκεκριμένο μήνυμα από τους Αφρικανούς ηγέτες για να σταματήσουν οι διακρίσεις κατά των ατόμων αυτών και βεβαίως όλες αυτές οι φρικτές ακρότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Κύριος Ιγνάνσιο Κοράο τώρα έχει τον λόγο ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Μαλάουι μαζί με άλλες αφρικανικές χώρες χαρακτηρίζεται από φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω προκαταλήψεων και απαράδεκτων πιστεύω του πληθυσμού. Συμμορίες ολόκληρες αλλά και μεμονωμένοι ε, στοχεύουν στην άσκηση βίας εις βάρος αυτών που υποφέρουν από αλφισμό και στερούνται φυσικά τις βασικές συνθήκες προστασίας. Ε, πρόκειται για φρικτά εγκλήματα, θα πρέπει να διώκονται οι, αυτοί που τα διαπράττουν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τις πολιτικές των μελών αυτών, έτσι ώστε να προστατευθούν με τη σειρά τους ε, αυτοί που ε, χαρακτηρίζονται από αλφισμό η δημιουργία σαν παράδειγμα ειδικών task force στις αστυνομικές δυνάμεις είναι κάτι το οποίο θα ήταν χρήσιμο νομίζω για τον πληθυσμό αυτό. Ευχαριστώ κύριε Κοράο. Ο κύριος Μποργέζιο έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το θέμα αυτό είναι ταμπού και ήταν ταμπού για πάρα πολλά χρόνια. Αρκετοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, θελήσαμε να καταθέσουμε ένα έγγραφο υπογραμμίζοντας ότι καταγγέλουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια το πρόβλημα αυτό ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς ήταν ταμπού. Ε, ποτέ δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά ε, με το θέμα αυτό. Είναι 27 οι χώρες στην Αφρική, ιδιαίτερα την υποσαχαρική Αφρική, που φύγονται από το πρόβλημα αυτό. Σε ορισμένες χώρες το πρόβλημα βέβαια είναι πολύ σοβαρό. Μιλάμε για το Μαλάουι, ο πρόεδρος Ματάρικα έχει καταγγείλει δημόσια την κατάσταση αυτή, αλλά δυστυχώς δεν έχουν ληφθεί μέτρα για να διωχθούν αυτοί οι οποίοι ε, χτυπούν ε, τους Αλμπίνους και ταυτόχρονα ε, επεξεργάζονται. Ε, είναι μια κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, που θα τη χαρακτήριζα δηλητηριώδη φρικτή. ιδιαίτερα όταν συζητάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αφρική, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να θέσει κι άλλο ένα ταμπού, το οποίο λίγοι θέτουμε, το θέμα του ρατσισμού εις βάρος των λευκών αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε ε, για τους ε, Αλβίνους ή κάτι το οποίο και αυτό στην ουσία οι διώξεις που υφίστανται εν πολλής είναι ρατσισμός εις βάρος αυτών που έχουν λευκή επιδευμίδα. Απαιτούνται λοιπόν συγκεκριμένες δράσεις. Η Ευρώπη θα πρέπει να ακουστεί πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνει μέχρι τώρα και η ίδια η Αφρικανική Ένωση θα πρέπει να μας ακούσει προσεκτικά και να αναλάβει πιέσεις, ε, να ξεκινήσει πιέσεις εις βάρος των μεμονωμένων κυβερνήσεων και να πάψει να καλύπτει τις ενέργειες αυτές οι οποίοι μας κάνουν όλους να ντρεπόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Μποργέζιο. Βέντα. Η κατάσταση των ανθρώπων αυτών είναι απαράδεκτη. Το ακούμε εδώ και χρόνια. Και πέρυσι, τον Ιούλιο, μας είχε απασχολήσει το θέμα. Δεν έχει υπάρξει όμως κάποια διαφοροποίηση. Δεν έχει υπάρξει προστασία των θυμάτων. Δεν έχουν υπάρξει μηχανισμοί που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους αυτούς να επανενταχθούν κοινωνικά. χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα τμήματα του σώματος τους για να παρασκευάζουν φαρμακευτικ... παρασκευάσματα φαρμακευτικού τύπου. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Όπως είπε και ο συνάδελφος του Νεκέλαμ η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της, του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας ζήτησε να ληφθούν κάποια μέτρα, κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα συμβεί απαιτείται να προστατευτεί επιτέλους η ομάδα αυτή και θα πρέπει οι οργανώσεις των πολιτών να παίξουν τον ρόλο που τους ανήκει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κιέγγε έχει το λόγο. Ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα του αλφισμού είναι ένα άγνωστο δράμα που όμως προκαλεί ε, εκατοντάδες θύματα στη διάρκεια των ετών και όμως πρόκειται για μια κληρονομική γενετική κατάσταση που αντίθετα θα έπρεπε να ε, καλύπτεται καταλήλως από τις υγειονομικές δομές της χώρας. Ε, κάποιες πρόοδοι έχουν επιτευθεί. πρώτα απ' όλα στην Τανζανία λόγω της ε, προς μεγάλης προσπάθειας ένταξης κάποια πράγματα γίνονται και χάρη στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα πρόγραμμα ε, δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, και της Αφρικανικής Ένωσης. Η πρωτα, ε, πρωταρχική ευθύνη κάθε κράτους είναι να προστατεύει τους ευαίσθητους ευάλωτους πολίτες του. Ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση του Μαλάι να αγγιηθεί η κατάλληλη προστασία στους ε, αλφικούς ώστε να προστατευτεί η ζωή τους και η προσωπική τους ασφαλή. Είναι απαράδεκτο αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι μόνο θύματα ακραίας βίας αλλά και θύματα δίωξης και κοινωνικού αποκλεισμού χρειάζεται μια πολιτιστική δράση που να θέσει τέλος στο στιγματισμό αυτών των ανθρώπων, από τα σχολεία να ξεκινά, ε, να εκκριζωθούν αυτές οι ε, παλιές πρακτικές που σήμερα το 2017 δεν θα πρέπει να έχουν χώρο σε κανένα χώρο παράδοσης. Οι ε, αλφικοί δεν πρέπει να εγκαταληφθούν στη μοίρα τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κέγκε. Ο κύριος Παουσπισίλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους ε, προλαλήσαντες. Είναι ε, θετικό το ότι θα εγκρίνουμε το ψήφισμα αυτό που καταδικάζει τις πρακτικές εις βάρος των αλφικών στην Αφρική. Είναι απολύτως σωστό το ότι περιγράφουμε λεπτομερώς όλα όσα αντιμετωπίζουν οι αλφικοί στην Αφρική, στο Μαλάουι συγκεκριμένα. Είναι πολύ περιγραφική λοιπόν αυτή η έκθεση και καλό θα ήταν η Κομισιόν ως το εκτελεστικό της Ένωσης να εστίαζε στην διπλωματία στην δυνατότητα να πιέσει αφρικανικές χώρες, το Μαλάουι εμπροκειμένο, για να προστατεύσει τον πληθυσμό των αλφικών. Το ψήφισμα αναφέρει επακριβώς ε, τις βιαιότητες που υφίστανται. Είναι απίστευτο ότι σημαίνουν αυτά τα πράγματα τον 21ο αιώνα και πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Σχέτμαν, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Η κατάσταση των αλφικών στην Αφρική είναι τρομακτική. Ε, μιλάμε για μεσαιωνικές ε, πρακτικές η δυσιδαιμονία ότι τα μέλη τους έχουν μαγικές δυνάμεις οδηγεί στο ότι πουλούν τα μέλη τους ε, για 75.000 δολάρια στη μαύρη αγορά. Οι άνθρωποι δηλαδή κινδυνεύει η ζωή τους. Και έχουμε συνεχώς περισσότερες δολοφονίες. Και συμβαίνει συχνότατα αυτό. αυτό πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα ενημέρωσης, διαφωτισμού για να καταλάβει ο κόσμος ότι ε, οι άνθρωποι δεν είναι φυλαχτά και ότι δεν έχουν ε, μαγικές δυνάμεις ε, στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα συστήματα εκπαίδευση και υγείας και βεβαίως ψυχολογική στήριξη. Επίσης συχνά ε, υπάρχουν, ε, σε κάποιες, υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις, αλλά δεν υπάρχει σοβαρή προστασία. Σας ευχαριστώ. Φαρέγκο για ένα λεπτό. Ο κύριος Φαρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, πριν από ένα χρόνο και πάνω ε, εγκρίναμε ένα ψήφισμα εδώ για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αλφισμό στην Αφρική, κυρίως και συγκεκριμένα στο Μαλάου. Ωστόσο, ε, στο Μαλάουι, στη Μοσαμβίκη, στη Νότια Αφρική και στη Τανζανία υπάρχει πρόβλημα και πολλά παιδιά ε, αλφικά πληρώνουν ε, αυτήν την, παρά, την, την παλιά παράδοση. Πολλοί πέφτουν θύματα εγκληματικών οργανώσεων και διακινητών. Είναι πολύ κερδοφόρο το εμπόριο αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορούμε παρά να καταδικάσουμε τη βία και τη διακρι... τις διακρίσεις κατά των ανθρώπων με αλφισμό και να θέσουμε, να βρούμε τους υπευθύνους και να στηρίξουμε όλες τις εξτρατείες ευαισθητοποίησης για και γνωστοποίηση αυτής της γενετικής ε, ε Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε αυτό το γενετικό apartheid. Ευχαριστώ Νικόλα. Ένα λεπτό. Νικόλα Σκαπούτο. Εκδιώκονται από τις κοινότητες τους, βασανίζονται. Γενικά η κατάσταση των ανθρώπων αυτών είναι απαράδεκτη σε πάρα πολλές από τις χώρες της υποσαχαρικής Αφρικής αλλά και στην Ινδία, σε ορισμένες περιοχές ε, κοντά στον Ινδικό ωκεανό πολλές φορές τμήματα των σωμάτων των νεκρών χρησιμοποιούνται για ιεροτελεστίες. Ε, η Amnesty International, η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει ότι είναι εκατοντάδες οι επιθέσεις αυτές και οδηγούν α, α, τους ανθρώπους αυτούς να ζουν μέσα στον τρόμο. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε όλες τις δυνατές δράσεις έτσι ώστε να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τις χώρες τις οποίες διαπιστώνονται τέτοιου είδους ενέργειες όπως το Μαλάουι να παρέχουν επιτέλους μια σωστή προστασία, να προστατεύσουν το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό. Υποστηρίζω το ψήφισμα το οποίο άλλωστε έχω συνυπογράψει τα άτομα με αλφισμό υφίστανται πραγματικές διώξεις πρόκειται για τουλάχιστον 20.000 συνανθρώπους μας δολοφονίες απαγωγές ακροτηριασμοί ταπεινωτικές συμπεριφορές είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν όχι μόνο στο μαλάουι αλλά σε αρκετές αφρικανικές χώρες. οι γυναίκες που γεννούν παιδιά με αλφισμό τα εγκαταλείπουν. όλα αυτά προέρχονται διότι υπάρχουν δυσιδαιμονίες υπάρχει η μαγεία και θεωρούν ότι τμήματα των μελών των ε, σωμάτων ε, των ε, αλφικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουν γιατροσόφια. αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση υπάρχουν κυνηγοί ατόμων με αλφισμό πρέπει να ποινικοποιηθεί η διακίνηση των ανθρωπίνων μελών και πρέπει να ενθαρρυνθεί η δράση σε τανζανία μοζαμβίκη νιγηρία και κένια να προχωρήσουν σε μέτρα για την προστασία των ατόμων που πάσχουν από αλφισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κέλλη, και εσείς για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ε, πραγματικά είναι αποτροπιαστική η κατάσταση των αλφικών στο Μαλάουι, την Τανζανία και αλλού. Το στίγμα, οι επιθέσεις και οι πωλήσει των μελών τους ε, είναι πραγματικά φρικιαστικά. Οι αλφικοί απομονώνονται, υφίστανται βία και παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Απευθύνω έκκληση στις ε, κυβερνήσεων χωρών να οδηγήσουν τους δράστες στην δικαιοσύνη γιατί φαίνεται ότι ε, απολαμβάνουν ε, ασυλίας αυτή τη στιγμή. Πρέπει επίσης να υπάρξει εκπαίδευση ε, για τους ανθρώπους αυτούς και στήριξη των θυμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υψώσει το αναστημά της για να μην συνεχιστούν αυτές οι παραβίασεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, να συγχαρώ τους ε, συναδέλφους ε, που θέλουν να σταματήσουν αυτές τις πρακτικές. Σας ευχαριστώ. Δεν ανώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι αυτοί οι οποίοι έχουν το χαρακτηριστικό αυτό ζουν ένα εφιάλτη. Αυτό ισχύει κυρίως στο Μαλάουι αλλά και λιγότερο σε άλλες χώρες της Αφρικής. Είναι λοιπόν ευθύνη των κρατών να λειτουργήσουν παιδαγωγικά προς τους πληθυσμούς τους αλλά να πάρουν και άμεσα μέτρα προστασίας γιατί ο πληθυσμός αυτός, οι κοινότητες αυτές δυστυχώς από τις δυσιδομονίες υποφέρουν όλο και περισσότερο. Πρέπει επίσης ε, να προστατεύσουμε και τις γυναίκες, διότι η δυσιδαιμονία λέει ότι η ερωτική ε, πράξη με ένα πρόσωπο που φέρει τον αλφισμό είναι κάτι το οποίο ε, προσφέρει πολλά. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, τα κορίτσια αυτά που δυστυχώς αντιμετωπίζονται φρικτά ήδη από την σχολική περίοδο. Είναι απαραίτητη η παρέμβαση των κυβερνήσεων, έτσι μόνο θα ξεπεραστεί ε, το πρόβλημα και έτσι θα προστατευθούν οι πληθυσμοί αυτοί. κύριος Πόλτσακ, τελευταίος ομιλητής, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι φρικτό το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα. Υπάρχουν δυστυχώς εκατοντάδες περιπτώσεις. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Δυστυχώς μιλάμε για τον 21ο αιώνα και όχι για το μεσαίωνα. Η παιδεία είναι ο τρόπος για να ξεραστούν οι προκαταλήψεις αυτές και οι δυσιδαιμονίες. Δεν είναι ο μόνος τρόπος όμως. Θεωρώ ότι απαιτείται να προστατευτεί η κοινότητα αυτή ε, το ταχύτερο δυνατόν. Πρέπει να υπάρξουν ποινές αυστηρότατες εις βάρος αυτών που τους κακό μεταχειρίζονται. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ε, προκαταλήψεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιούροβα εξ ονόματος της κυρίας Μογκερίνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε την δυνατότητα να πάρω μέρος σε ένα σημαντικό θέμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει δυστυχώς μια χειροτέρευση στο θέμα της αντιμετώπισης των Αλμπίνων στο Μαλάουι και σε άλλες χώρες της περιοχής. Υπάρχουν πολλαπλές μορφές διάκρισης της σβάρους ε, τους, υπάρχει εμπορία ανθρωπίνων μελών και φυσικά προηγούνται δολοφονίες. Ε, είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί επανειλημμένα και εδώ και γι' αυτό θα πρέπει να αναλυφθούν επιτέλους πρωτοβουλίες και δράσεις. Δράσεις οι οποίες έχουν προταθεί στο παρελθόν και προτάσσονται επίσης και σήμερα. Εμείς ε, έχουμε ζητήσει από τις χώρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό επιγόντως να λάβουν μέτρα υπέρ ε, το, της κοινότητας αυτής και ταυτόχρονα να τιμωρούνται ε, από την δικαιοσύνη αυτή που διαπράττουν αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες. Απαιτείται συνεργασία και διασυνοριακή επίσης γιατί πάρα πολύ συχνά το θέμα αυτό έχει περιφερειακή διάσταση. Ταυτόχρονα έχουμε υποστηρίξει ε, και την ανάγκη να καταπολεμηθεί το στίγμα εις βάρος των Αλμπίνων και ταυτόχρονα έχουμε ζητήσει οι ανάγκες τις οποίες έχουν ε, στον τομέα της παιδείας, στον κοινωνικό τομέα, στον ιατρικό τομέα να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να βοηθήσουμε και την κοινωνία των πολιτών η οποία και αυτή παίζει σημαντικό ρόλο στο να αντιμετωπιστούν οι προκαταλήψεις και οι δυσιδαιμονίες η διεθνής κοινότητα όλο και περισσότερο κινητοποιείται σε σχέση με το πρόβλημα αυτό. Ε, στις 7 Ιουνίου ήταν η ημέρα για την αναγνώριση του προβλήματος των ε, Αλμπίνο. Ε, πρέπει λοιπόν, έχουμε ζητήσει να υπάρξει μάλλον και μία έκθεση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τα ανθρώπινα δικαιώματα της συγκεκριμένης αυτής κοινότητας και οι κυβερνήσεις δείχνουν ότι αρχίζουν να ανησυχούν για, για το μέγεθος του προβλήματος αυτού, για την κλίμακα του προβλήματος αυτού. Είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Εμείς μέσω των αντιπροσωπιών μας στις διάφορες χώρες συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος μας είναι οι, αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν το θέμα του αλφισμού να προστατεύονται από τις διακρίσεις και από τη βία. Ευχαριστώ την Επίτροπο Γιούροβα, ευχαριστώ όσους πήραν το λόγο. Έχω λάβει οκτώ προτάσεις ψηφίσματος καταληκτικές της συζήτησης. Ε, τελείωσε η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει